Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Το 12ο σημείο της ημερησίας διάταξης, δημοκρατικός έλεγχος του προγραμματισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ανάπτυξη. Αυτό αποσύρθηκε από την ημερησία διάταξη όπως ανακοινώσαμε στην αρχή της συνεδρίασης. Σημείο 13. Πρωτοβουλία για μια αποτελεσματική εταιρική σχέση στον τομέα της ανάπτυξης διαθρωμένος διάλογος για μια αποτελεσματική εταιρική σχέση στο τομέα της ανάπτυξης. Ξεκίνησε επισήμως το Μάρτιο του 2010 με ανακοίνωση του Επιτρόπου κ. Πίλμπαλξ. Συγκεκριμένα, ο διαθρωμένος διάλογος προσπαθεί να βρει μέσα μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική την εταιρική σχέση και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ενδιαφέρονται για αυτό. 2 με 4 Ιουνίου θα υπάρξει το πρώτο περιφερειακό σεμινάριο στο Μπαμακό. Ο συνάδελφος ο κύριος Νόισερ συμμετείχε στο σεμινάριο και θα ήθελε να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια από την Επιτροπή ο κύριος Μπαλιό θα μας ενημερώσει για τα επόμενα περιφερειακά σεμινάρια καθώς και για αποτελέσματα που αναμένουμε από αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Νόισερ, 15 λεπτά το μέγιστο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω και εγώ ότι ο διαρθρωμένος διάλογος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και γι' αυτό θα σας αναφέρω εν συντομία τα πεπραγμένα του πρώτου περιφερειακού συνεδρίου που έλαβε χώρα στον Παμακό στο Μάλι. Η Κομισιόν έχει ήδη διοργανώσει ε, μια σειρά από τέτοια σεμινάρια σε σχέση με το διαρθρωμένο διάλογο. Το πρώτο, όπως ελέγχθη, ήταν στο Μάλι, στο Παμάκο. Ο στόχος αυτών των διαλόγων είναι η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές αρχές να συμμετάσχουν καλύτερα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας για την ανάπτυξη που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι οι νέες διαδικασίες βοήθειας όπως είναι ο, η βοήθεια, η αρρωγή προς τον προϋπολογισμό και η τομεακή βοήθεια προς τον προϋπολογισμό. Στο Μπαμάκο ασχοληθήκαμε με τα θέματα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και την τελευταία μέρα του σεμιναρίου για τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Η Επιτροπή Ανάπτυξης είχε ήδη εμπλακεί από την αρχή της διαδικασίας αυτής του διαρθρωμένου διαλόγου, ο κύριος Γκέρνς, πρόεδρος ομάδας εργασίας 4, στην οποία τα προγράμματα που αφορούν μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τοπικές αρχές εξετάστηκαν, έλαβε μέρος σε αυτό το τμήμα του διαλόγου και επίσης η γραμματεία της Επιτροπής μας ήταν παρούσα στην ε, διαδικασία αυτή και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Βαλέρια για την πολύ καλή της υποστήριξη. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η ενεργή εμπλοκή του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική για την ε, επιτυχία αυτού του εγχειρήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας από τους κύριους μέσα σε εισαγωγικά παίκτες για τα θέματα αυτά και μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο για τη συνεργασία εθνικών κοινοβουλίων, τοπικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το κοινοβούλιο μας μπορεί λοιπόν να είναι και ο εκπρόσωπος της συνεργασίας αυτής και να εμπλέξει τα Εθνικά Κοινοβούλια, την Κοινωνία των Πολιτών και τις τοπικές αρχές που μπορούν να είναι πραγματικά ένα σημαντικό επόπτης για την ορθή εφαρμογή των νέων αυτών τρόπων υποστήριξης, συγκεκριμένα της αρρωγής προς τον προπολογισμό και της συμμετοχής της τομεακής υποστήριξης προς τον προπολογισμό. Όλα τα έγγραφα αυτά είναι βέβαια στα αγγλικά, είναι κάπως δύσκολο στα γερμανικά να τα μεταφράσει όλα αυτά κανείς και υπάρχουν και πολλές τεχνικές έννοιες τις οποίες δυσκολεύουμε να τις περάσω στα γερμανικά. Το πρώτο τμήμα λοιπόν του σεμιναρίου αφορούσε την κοινωνία των πολιτών. Το πρώτο τμήμα του σεμιναρίου αφορούσε την παρουσία των τοπικών αρχών και των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Ευρώπη και την Αφρική. Το σεμινάριο υπήρξε μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία βορρά-νότου και νότου-νότου μεταξύ τοπικών αρχών και μη κυβερνητικών φορέων. Υπήρχαν πάνω από 50 φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 30 εκπρόσωποι τοπικών αρχών από τις χώρες εταίρες που συμμετέσχαν σε αυτό το σεμινάριο και κατά την άποψή μου ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών και συνεργασία μεταξύ ομοτήμων. Η Κομισιόν οργάνωσε μια σειρά από σεμινάρια που θα εστιάσουν στα εξή θέματα. Ρόλος και προσθέμενη αξία της κοινωνίας των, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών και των τοπικών αρχών μέσα στη διαδικασία ανάπτυξης. συμπληρωματικό ρόλο και συνεκτικότητα τη δράση των εταίρων αυτών για συνεργασία και μηχανισμός μηχανισμός αποτίμησης της προσθέμενης αξίας της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει επίσης να υπάρξει και περισσότερη εστίαση στο ρόλο των εμπλεκομένων και τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα βελτιώσει τον διάλογο μεταξύ τοπικών εμπλεκομένων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών από την Ευρωπαϊκή και την Αφρικανική πλευρά, ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και την πρόκληση της τοπικής διακυβέρνησης στην Αφρική και επίσης βελτιώσεις στο μηχανισμό αυτό, ένα σύστημα υποβολής προτάσεων, ταυτοποίηση διαφορετικών μηχανισμών παράδοσης βοήθειας, ώστε να αντανακλάται και η πολυμορφία των εμπλεκομένων. Το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου αφορούσε τις τοπικές αρχές. Η Κομισιόν παρουσίασε τις κύριες δραστηριότητες σε σχέση με το ρόλο των τοπικών αρχών. Με επομένως στόχο να προωθήσει τη αποκεντρωμένες αυτές επαφές με παρουσία της Κομισιόν και, το, και της Επιτροπής των Περιφερειών, μέσα στα πλαίσια των οποίων μπορούν να έρθουν σε συνάντηση οι εκπρόσωποι από την ευρωπαϊκή πλευρά και την αφρικανική πλευρά των τοπικών αρχών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2011. Η διαποκεντρωμένη αυτή συνεργασία λοιπόν θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα ιονί οδικό χάρτη των πρωτοβουλειών των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών για την ανάπτυξη και συνεργασία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συντεριάσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες με τις ανάγκες της επιτόπιας, ώστε να ενισχυθούν και οι σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρες. Τέλος, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών από τρεις αφρικανικές χώρες παρουσίασαν τρία καινοτόμα σχέδια. Η απογευματινή συνεδρίαση εστίασε και πάλι στο ρόλο των τοπικών αρχών και την ικανότητά τους να δημιουργήσουν εταιρικέ σχέσεις και καινοτομία στην χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. Υπήρξαν κάποιες συστάσεις από τη δική μας πλευρά. Καταρχήν, να υπάρξει μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τοπικών αρχών και μη κυβερνητικών φορέων που να είναι πιο διαρθρωμένοι <clears throat> στην ε, φάση προγραμματισμού και αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο. Η διαβούλευση μεταξύ των φορέων αυτών θα πρέπει να έχει σαν στόχο να αναπτύξει ένα σταθερό και επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών και των τοπικών αρχών. Δεύτερον, μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητέ μα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ικανότητα των τοπικών αρχών και των οργανώσεων βάση τη κοινωνία των πολιτών. Τρίτον, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών θα πρέπει να λάβει χώρα και να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανότητα. Τέταρτον, τέταρτο, οι τοπικέ αρχέ θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία και το συντονισμό των δράσεών του με άλλου εμπλεκομένου. Θα πρέπει να ενισχύσουν λοιπόν και τη συμμαχία του με εθνικά κοινοβούλια και άλλου εμπλεκομένου. μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι οι οργανώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης ζητούν να υπάρξει καλύτερος ε, διάλογος με συντονιστές της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέμπτον, θέλουμε να δώσουμε υποστήριξη για την αποκέντρωση τόσο σε εθνικό επίπεδο, τόσο επίσης και σε θεσμικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο. Έξι σε σχέση με τους τρόπους χρηματοδότησης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την πολυμορφία τους και ζητούν να υπάρξει χρηματοδότηση που να αντανακλά την πολυμορφία τους, επομένως να υπάρξουν καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Τονίζουν αυτές οι οργανώσεις ότι ο μηχανισμός υποβολής προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ειδική ποσόστοση για οργανώσεις βάσης. Εύθομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένας από τους κύριους παίκτες στον διαρθρωμένο αυτό διάλογο και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντική και η συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες αυτές τις φάσεις θα πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Η συνάντηση εργασία στι Βρυξέλλες και τα περιφερειακά σεμινάρια έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα λοιπόν σα ενθαρρύνω να συμμετάσχετε στην επόμενη σύνοδο εργασία στι Βρυξέλλε στι 12 Ιουλίου. Τέλος, επειδή έχουμε κάποιους εκπρόσωπους από πλατφόρμες μη κυβερνητικών οργανώσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να τους προσκαλέσω όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στον διαδρομένο διάλογο στη μελλοντική αυτή συνεδρίαση ad hoc για να μπορέσουμε να έχουμε διάλογο η Επιτροπή μας με τους εκπροσώπους αυτών των πλατεφορμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαλιό. Έχετε το λόγο για 10 λεπτάκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Μέσνερ για την έκθεσή του σχετικά με αυτά που έζησε στον Παμακό. Υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες πτυχές στα συμπεράσματά του και θα υπάρξουν και αρκετά σχόλια. Αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπήκε σε μια διαδικασία διαρθρωμένη αρκετά μακρόχρονη, θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, όμως αυτός ο περιορισμός ο χρονικός με ένα πρόγραμμα εργασίας αρκετά λεπτομερές θα μας επιτρέψει στο τέλος της διαδικασίας, στο τελικό σεμινάριο επί Ουγγρικής Προεδρίας τον επόμενο Μάιο να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία. Είχαμε και την εμπειρία της διαδικασίας του Παλέρμου. Τότε ουσιαστικά επρόκειτο απλά για συζήτηση με τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τον τρόπο χρήσης ε, των ε, χρηματοδοτικών ε, μέσων που ήταν διαθέσιμα σε αυτούς. Τώρα, η χρηματοδότηση προς τις ε, μη καπαόμικρον στο παρελθόν αφορούσε κυρίως τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο νέος κανονισμός όμως αύξησε σημαντικά και άνοιξε σημαντικά την δυνατότητα συμμετοχής σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις ενδιαφερόμενες χώρες. Δεν θέλουμε βεβαίως να αντιπαραθέσουμε κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, όμως η έννοια της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ πιο δυναμική. Μας επιτρέπει λοιπόν να έχουμε συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας στην ανάπτυξη. Αυτή είναι η θετική πλευρά των πραγμάτων. Είναι αλήθεια ότι η Κομισιόν πριν ξεκινήσει τη διαδικασία είχε υποστηπιέσεις ε, κυρίως από το Κοινοβούλιο. Θα θυμάστε και την ε, συνεδρίαση της Κοκομπού τον προηγούμενο Οκτώβριο με τον Γενικό Διευθύντη τον κύριο Ρισελ όπου παρουσιάστηκαν ε, τα αποτελέσματα για τους λογαριασμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μη φορέων και των διαδρομών χρηματοδότησής τους τότε μία διαπίστωση ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με μη κρατικούς φορείς, όμως πρόκειται κυρίως για δραστηριότητες ad hoc, διάλογο ή οτιδήποτε άλλο, που πάντα στρέφονταν γύρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς μπορεί να εφαρμόσει αυτό, πώς μπορεί να βελτιωθεί κάτι άλλο, ποια θα έπρεπε να είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το σύστημα παροχής βοήθειας. Και βεβαίως υπήρχε και το σύστημα διαλόγου πέρα από τις τεχνικές συζητήσεις που αφορούσε το ρόλο κάθε φορέα. Άρα, τώρα ο στόχος αυτού του διαθρωμένου διαλόγου είναι να διαπιστώσουμε πώς κάθε φορέας μπορεί να βελτιώσει την αποδοσή του, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά του μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας ε, πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Έχουμε κάνει πολλά θετικά, όμως πρέπει να δούμε κάτι περισσότερο. Παρόλο που σε ορισμένες χώρες μας όντως βοήθησε η δραστηριότητά μας στο να περάσουμε από την απόλυτη φτώχεια σε κάποια μεγαλύτερη, καλύτερη φάση εφημερίας. Μέσω του διαρθρωμένου διάλογου ψάχνουμε να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε περισσότερο τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στις εταιρικές χώρες. Μιλάμε λοιπόν για διάφορες πλατφόρμες, για διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ένας τρόπος να το επιτύχουμε είναι να ανοίξουμε το διάλογο με τις οργανώσεις αυτές του Νότου και να μάθουμε τα αιτήματά τους. Για αυτό το λόγο η διαδικασία λαμβάνει χώρα εναλλάξε στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της ομάδας Α, όπου έχουμε και τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών και να αλλάξει πάλι έχουμε τα τοπικά σεμινάρια που θα είναι τέσσερα. Ένα έγινε ήδη στις αρχές Ιουνίου στο Μακό, θα υπάρξει άλλο ένα στις 14 Σεπτεμβρίου στο στη Νότιο Αμερική. Μετά θα έχουμε το σεμινάριο για την Ασία το Νοέμβριο με περίπου 15 χώρες ε, της ε, Ασίας και θα καταλήξουμε με τις ε, γειτονικές χώρες. Άρα, κάθε φορά που έχουμε ένα σεμινάριο, το σεμινάριο διορίζει κάποιους εκπροσώπους των χωρών για να έρθουν στις Βρυξέλλες. Έτσι τον Ιούλιο θα έχουμε 8 εκπροσώπους της Αφρικής, τρεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τρεις των τοπικών αρχών και οι οχτώ θα είναι της κοινωνίας των πολιτών. Αυτοί θα συμμετέχουν στις εργασίες μας τις Βρυξέλλες με στόχο να έχουμε έναν ισορροπημένο διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου να συνεχίσει να στηρίζει αυτή τη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά. Βεβαίως δεν πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης, απλά για διαδικασία διαλόγου. Όμως το στίχημα για την Επιτροπή είναι ότι έχοντας λάβει τις πληροφορίες, έχοντας κάνει αυτό τον διαλόγο, όλες αυτές οι οργανώσεις ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών, ε, οι τοπικοί φορείς, αλλά και εμείς ως Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες γνώσεις και να τις μετασχηματίσουμε σε προτάσεις για ένα νέο τρόπο συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, να πω ότι αυτό αφορά όλη την εξωτερική συνεργασία, όχι μόνο π.χ. τα θεματικά προγράμματα. Αφορά όλη τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στα πλαίσια των εξωτερικών προγραμμάτων και της δικής μας κοινωνίας των πολιτών, αλλά κυρίως της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες του Νότου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει το λόγο. Έχω εγώ ένα ερώτημα βέβαιος. Υποθέτω ότι τα αιτήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια στις γραμμές του προϋπολογισμού. Πώς αποφασίζετε ποιος θα λάβει τη χρηματοδότηση και ποιος όχι. Κάθε χρόνο πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί περίπου ένα δισεκατομμύριο, δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 10 με 13% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Γενικά λοιπόν, αυτό γίνεται μέσω προσκλήσεων για εκδήλωση προτάσεων. Δεν είναι ότι αποφασίζει η Κομισιόν πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οι κανόνες για την υποβολή προτάσεων και στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση της σχετικότητας κάθε σχεδίου, της αξία του και επομένω αποφασίζεται η χρηματοδότησή του το πρόβλημα που συμβαίνει, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, είναι ότι είμαστε λίγο θύματα της επιτυχίας μας εννοώ. Και για κάθε πρόσκληση δεχόμαστε χιλιάδες προτάσεις, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στις τοπικές αντιπροσωπείες μας. Ως εκ τούτου, κατά μέσον όρο, μόνο 5% των προτάσεων τη χάνουν χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει τεράστιο όγκο εργασίας και στις Βρυξέλλες, αλλά και στις ε, αποκεντρωμένες οργανώσεις. Αυτό λοιπόν είναι και αντικείμενο συζητήσεων που κάνουμε τώρα με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό το οποίο θα αντιμετώπιζε καλύτερα αυτές τις προκλήσεις. Χωρίς να θέλουμε να απορρίψουμε το βρέφος μας με τα ύδατα κολύμβησης αυτού του ιδίου του βρέφους, θέλουμε να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Α, ο κύριος Ντέβας. Πρώτα, έχετε το λόγο, κύριε Ντέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσε ότι, άκουσα ότι πρέπει να διεκπαιρεώσει χιλιάδες προτάσεις. Πόσες ανθρωπόρες λοιπόν δαπανάτε και στην Κομισιόν αναλύοντας και επεξεργαζόμενοι χιλιάδες προτάσεις και πόσος χρόνος και ανθρωπόρες δαπανώνται παρακολουθώντας τις προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί. Σίγουρα, πολύ, υπερβολικά πολύ χρόνο ε, με την επεξεργασία χάνουμε και όχι αρκετό με την παρακολούθηση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα των, του κανονισμού, του δημοσιονομικού κανονισμού, που σε κάποιο βαθμό ορίζει την ε, πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ως το σύστημα όσο το γενικό ισχύον σύστημα. Εμείς ε, προφανώς έχουμε μια πιθανή εναλλακτική, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται μόνο κατ' εξαίρεση. Όσον αφορά τις ε, ανθρωπόρες, ε, θα μπορώ βέβαια να σας δώσω τώρα πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αρχίζουμε με ένα σημείωμα σύλληψη, μετά έχουμε την πλήρη πρόταση, μετά γίνονται επιτροπέ εκτίμηση αξιολόγηση με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αλλά και με συναδέλφους από όλε τις αντιπροσωπείες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση. Και τέλος βγαίνει, μετά από όλα αυτά βγαίνει η τελική απόφαση. Όντω θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσες, πόσες ώρες δαπανούμε. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να γίνει μια εκτίμηση. Ωστόσο, ορισμένες ε, προσκλήσει είναι πιο εύκολες από άλλες. Μπορείτε να τα μεταδιαβιβάσετε όλα αυτά στον Επίτροπο ή μήπως θέλετε να του θέσω ερώτηση στην Ολομέλεια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να διαβιβάσω την ερώτηση και να απαντήσω και γραπτός, είτε στην Ολομέλη είτε ε, γραπτός. Κύριε Νόιζερ, έχετε το λόγο για να ε, ολοκληρώσετε. Κυρία Πρόεδρε, για να κλείσω, πρέπει να σας κάνω την εξής παρατήρηση. Χθε σε ένα σημείο της ημέρησης διάταξης συζητήσαμε για την εποπτεία σε ό,τι αφορά τις αρρωγές στον προϋπολογισμό. Και είπαμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των κοινοβουλίων στα αναπτυσσόμενα κράτη και να υπάρξει επίσης και η δυνατότητα της ε, επιφόρτισης των ελεκτικών συνεδρίων με τον έλεγχο αυτής της ε, αρρωγής στον προϋπολογισμό. Όταν όμως έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, τότε είναι ένα κοινοβούλιο μονάχα το οποίο μπορεί να ελέγξει αυτή την κυβέρνηση, αλλά πολύ συχνά και το ίδιο αυτό το κοινοβούλιο είναι διεφθαρμένο ή ακόμα πιο διεφθαρμένο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπίσουν αυτή την διαφθορά. Γι' αυτό λοιπόν σημαντικό να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές και στις χώρες του Νότου. Γι' αυτό η έκκλησή μου, εγώ τονίζω και πάλι, ότι θα ήταν σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότερο κοινοβουλευτικοί να συμμετέχουν σε αυτή τη δομή του διαρθρωμένου διαλόγου, ώστε να υπάρχει όρο και μεγαλύτερη επιρροή τη ε, δική μα πλευρά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει 14ο σημείο της ημέρησης διάταξης μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικοψαρευτικής πολιτικής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νήσων του Σολομόντος. Ο κύριος Ντέβα είναι ο εισηγητής επί τη βάση της εντολής που δόθηκε στην Κομισιόν από το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νήση Σολομόντος στις 17 Σεπτεμβρίου του 2009 μονογράφησαν μια συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα για τρία χρόνια στον τομέα της αλίας. Αυτό επιτρέπει στην, στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψαρεύουν στα νερά του νήσων Σολομόντος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και η συνεργασία των δύο πλευρών και προωθείται ένα πλαίσιο εταιρική σχέσης που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας πολιτικής αλίας και μιας αηφόρου εκμετάλλευσης των ηχθείων των νήσων του Σολομόντος και από τις δύο πλευρές. Η Επιτροπή Αλληλείας είναι η αρμόδια για γνωμοδότηση στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Αλίας προβλέπει στις 30 Αυγούστου να δοθεί αυτή η γνωμοδότηση. Εμείς λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε τη δική μας πρόταση στη συνεδρίασή μας 12 και 13 η Ιουλίου. Κάνουμε σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντέβαν, ο οποίος είναι εισηγητής, ο οποίος έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πάμε πολύ μακριά ως τις του Σολομόντος, εάν θέλουμε να ψαρέψουμε εκεί. Ούτως ή άλλως όμως η Συμφωνία Ευρωπαϊκής ευρωπαικης ενωση και Νήσων Σολομόντος εξέπνευσε τον προηγούμενο Οκτώβριο το νέο πρωτόκολλο ισχύει από τις 9 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά από τις συνθήκες Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να δώσει σύμφωνη γνώμη ή να αρνηθεί να δώσει σύμφωνη γνώμη βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 και του άρθρου 118 παράγραφος 6α των συνδικών σε σχέση με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δίνει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερη επιρροή στις αλληλευτικές συμφωνίες. Πρέπει να θυμηθούμε επίση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να εφαρμόζεται προσωρινά, χωρί την έγκριση του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η έγκριση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ψηφιστεί κυρίω από την Επιτροπή Αλίες η οποία θα τύχει τη γνωμοδότησή μα πριν από το τέλο Αυγούστου, η δυνατότητα άρνηση τη έγκριση θα πρέπει να συνάδει με τις εξή προϋποθέσεις. Πρώτον, η διαφάνεια της διαδικασίας για τον εντοπισμό των συνολικών αλλιευμάτων θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση του μηχανισμού σε σχέση με την διαφθορά, την ενδεχόμενη διαφθορά που μπορεί να είναι θέμα στην χώρα αυτό. Και οι νήσοι Σολομόντο φαίνεται ότι είναι από τις πιο διεφθαρμένε χώρες του κόσμου, επίση και οι ηχθείς του. Και τρίτον, μια ρήτρα για τις τοπικές κοινότητε που να εξασφαλίσει την καλύτερη διαβίωση των τοπικών αλλιέων. <clears throat> για τι λεπτομέρειε, επειδή μερικέ φορές είναι πολύ εντυπωσιακά τα πράγματα αυτά, θέτει ένα όριο για την αλίευση τόνου. και η Συμφωνία για την αλλιεύση Τόνου έχει ένα όριο 4.000 τόνων. Τόνου. Αυτό όμως δεν περιορίζει τα αλλιεύματα σε 4.000 τόνους τόνων. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει σε, μέσα σε αυτό το όριο 65 ευρώ ανατόνο τόνου. Αν συλλέξουν περισσότερους τόνους από 4.000 τόνους τόνων, αλλιεύουν αυτά τα αλλιεύματα, αλλά πληρώνουν περισσότερο. Επομένως έχουμε μια συμφωνία με όριο 4.000 τόνους και στην περίπτωση που αλλιεύσουμε περισσότερους τόνους θα τους δώσουμε περισσότερα λεφτά. Αλλά οι νήσεις Σολομόντος δεν έχουν ιδέα πόσους τόνους θα αλλιεύσουμε. Θα πρέπει να βασιστούν στη δική μας διάκριση για το πόσους θα αλλιεύσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει οι αλλοί της Ευρωπαϊκή Ένωση να πούνε στις νήσους Σολομόντος πιάσαμε τόσους και επειδή πιάσαμε τόσους θα σας πληρώσουμε. Βέβαια αργότερα θα σας πληρώσουμε. Μπορείτε να το φανταστείτε να μπλέκεστε σε μια τέτοια συμφωνία στην Ευρώπη. Όχι. Λοιπόν. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κάτι ακόμα. Ένα ακόμα στοιχείο πρέπει να λάβουμε υπόψη αν είναι διπλάσια η αλίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσουν αργότερα. Α πούμε, αν φτάσουμε σε 9.000 τόνου. τότε θα πληρώσουμε για 8.000 τόνου, αλλά για, το τελευταίο, για τους τελευταίους τόνους η χώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον επόμενο χρόνο για να πάρει τα λεφτά της. Μην με ρωτάτε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει παροχή εκθέσεων, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος του τι αλλιεύεται, οι αρχέ του Σολομόντος δεν θα έχουν κανένα επόπτη στα πλοία, οι αλληλεί μας θα πούνε τόσα πιάσαμε, γεια σα. όσα έρθουν και όσα πάνε. Και γεια σα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δίκαιο προς τις νήσους του Σολομόντος. Και χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ παρούσα και η πρόεδρός μας και θα είναι στην αλληλευτική ακρόαση για να μπορέσει να παρουσιάσει την άποψή τη. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξή. Οι νήσοι Σολομόντο έχουν συμφωνήσει για μια περιφερειακή προσέγγιση στα, στις διεθνείς συμφωνίες, δηλαδή έχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν τις συμφωνίες όλων των χωρών της περιοχής έναντι συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τηρούνται αυτά τα συμπεφωνημένα. Απάντηση. Δεν ξέρουμε. Πώς επαληθεύουν τα αλλιεύματα οι αρχές των νήσων Σολομώντος που βρίσκεται σε θέση 111 από 180 σε ό,τι αφορά την συνολική διαφορά ποιος επαληθεύει τα συνολικά αλλιεύματα ένας ανεξάρτητος φορέας ή κάποιος ο οποίος δίνει μπαχτσίσει μερικά εκατοντά, μερικές εκατοντάδες δολάρια σε κάποιον υπάλληλο. Και επίσης πόσα από τα χρήματα που δίνονται στην κυβέρνηση θα χρησιμοποιηθούν για τους στόχους ανάπτυξης των φτωχοτέρων στις νήσους Σολομόντος, μεταξύ των οποίων και οι αλίες, για να βελτιωθεί η κατάρτισή τους στο βιωτικό τους επίπεδο κτλ. Πρόκειται για βιοτεχνική αλληλεία, η οποία βρίσκεται σε πολύ μειονεκτική θέση όταν έχονται μεγάλα πλοία, το είναι στη Σενεγάλη, πολλοί έχουν, έχουν σκοτωθεί όταν τους χτύπησαν μεγάλα αλλιευτικά πλοία κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια άκρα επιφυλακτικότητα σε σχέση με όλα αυτά και να προχωρήσουμε να έχουμε και κάποια εξάρτηση από την παροχή εγγυήσεων για να δώσουμε την έγκρισή μας. Αν δεν έχουμε λοιπόν εξάρτηση και διαφάνεια και παροχή εκθέσεων δεν πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Βέβαια αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Αλίας και θέμα ημών με ύψιλον, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία. η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συμφωνία. Εγώ ως δεν ξέρω από τιμέ. 60 ανατόνο τόνου που είναι ήδη είδος ε, απειλούμενο, είναι φυσιολογική αυτή η τιμή όχι. Δεύτερον, είπατε ότι θα θέσετε προϋποθέσεις για την έγκριση της συμφωνίας. Επειδή όμως ε, ουσιαστικά ήδη εφαρμόζεται και εμείς απλά την εγκρίνουμε, αν υπάρξουν εκ των υστέρων ε, αλλαγές. Υπάρχει δυνατότητα να περάσουν οι αλλαγές μας και να εγκριθούν ή όχι. Ή απλά πρέπει να πούμε ναι ή όχι και ενδεχομένως να είναι καλύτερο να πούμε όχι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου λοιπόν για τις τιμές και για το αν είναι δυνατές αλλαγές. Να απαντήσω κυρία Πρόεδρε. Το ποσό που πληρώνουμε στα νησιά Σολομόντα είναι 216.000 ευρώ για 4.000 τόνους. Θεωρώ ότι ένα κιλό τόνου στο ψαράδικο της γειτονιάς κάνει 35, κιλό, 35 ευρώ, με 35 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αν είναι προέλευση νησιών Σολομόντα ή όχι. Αλλά ένα τόνο τόνου λιανική τιμή 35.000 ευρώ. Εμείς πληρώνουμε 65 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης. Πληρώνουμε 65 ευρώ τον τόνο και δεν ελέγχονται καν. Και μιλάμε για λιανική τιμή 35.000 ευρώ για αυτόν τον τόνο. Θεέ μου πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις τροπολογίες, πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Άρα πρέπει να έχουμε πολύ καλούς λόγους για να πούμε όχι. Σιγά σιγά όμως τους βρίσκω. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Συζητάμε μια πολύ συγκεκριμένη αλλιευτική συμφωνία που αφορά τα νησιά του Σολομόντα μόνο. Όμως πρέπει να συζητήσουμε και συζητάμε στην Επιτροπή μας όλες τις ε, FPAs ε, γιατί νομίζω ότι τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στις υπόλοιπες δεν υπάρχει συνοχή. Άρα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να επιδοτούμε μεν την αλία μας αλλά χωρίς να προκύπτει ασυνάφεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Να πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία με τα νησιά αυτά υπάρχουν βελτιώσεις, όμως ε, υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Ναι, μεν υπάρχουν ρυθμίσεις όσον αφορά την παράνομη άναρχη αλία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αρκεί. Και βεβαίως όταν βλέπουμε ότι ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να παρακολουθούμε την άναρχη αλία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης να πω ότι αυτή η συμφωνία έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2009. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε κάτι που ήδη εφαρμόζεται. Να πω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι πολύ επιφυλακτική στη γνωμοδότησή της. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μία νέα προσέγγιση για τις ε, συμφωνίες τις αλλιευτικές. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιες συμφωνίες για τις χώρες που εξάγουν ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί υπάρχει συνεργασία των Γενικών Διευθύνσεων Εμπορίου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που συμπεριλαμβάνουν μέτρα για τη διαφάνεια και την συμμετοχή της ε, κοινωνίας. Εδώ όμως στις αλληλευτικές συμφωνίες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό. Μας ενδιαφέρουν απλά τα αλληλευτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για τη διαχείριση των αλληλευτικών συμφωνιών και πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να την ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής. κυρία Κέλλερ, κάτι ακόμη, ένα ερώτημα επί της ουσίας και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αρσένη. Αν είπατε, αν κατάλαβα καλά, μετά τις 4.000 τόνους πρέπει να πληρώσουν επιπλέον πληρώνουν και περισσότερα ανατόνο ή την ίδια τιμή ανατόνο. Ο κύριος Δέβα, την ίδια τιμή και αργότερα. Και αν τα λεύματα είναι περισσότερα από το διπλάσιο, πολύ πιο αργά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, τι νόημα έχει αυτό, αφού δεν γνωρίζουμε πόσα είναι τα λιεύματα στην πραγματικότητα. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο για να συνοψίσετε εφόσον δεν έχουμε εκπρόσωπο της Επιτροπής. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αφού το εξέτασα όλο αυτό, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, έχω σοκαριστεί. Λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για τους στόχου, θέλουμε να εκριζώσουμε τη φτώχεια, μα κάποιοι από τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι αλληλείς. Ζουν σε αλληλευτικές περιοχές, τα νησιά του Σολομόντα, Δεν πρόκειται να, και για κόσμος που εκεί δεν πρόκειται να αφαιρεθεί από οτιδήποτε και αν κάνουμε εμείς εδώ. Οπότε τουλάχιστον θα έπρεπε να φτάνουν εκεί αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για 260.000 ευρώ για 4.000 τόνους. Δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα θα τα δουν οι ψαράδες και πόσα βλέπει, βλέπει ο υπουργό ή η κυβέρνηση. Οπότε ολόκληρη αυτή η υπόθεση της αλληλείας θα πρέπει να εξεταστεί από την ε, οπτική της ανάπτυξης. Εγώ εύχομαι καλή τύχη στον Πρόεδρο σήμερα στην αγώνα, στην ακρόαση που θα γίνει με την Επιτροπή Αλίες. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Να σας δώσω τις ημερομηνίε για τις επόμενες μας συνεδριάσεις ε, στις Βρυξέλλες 12 ε, Ιουλίου 3 με 6.30 και 3η 13 Ιουλίου από τις 9 μέχρι τις 5.30. Να σας θυμίσω πως το απόγευμα γίνεται η κοινή ακρόαση της Επιτροπής Αλληλείας και Ανάπτυξης για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αυτή η ακρόαση θα γίνει στο ΠΑΣΕΣ στην 5B001 αίθουσα και ελπίζω πως θα έρθετε όλοι. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν.